Καλησπέρα, συνάδελφοι. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση. Πρώτο θέμα. Δήλωση της Επιτροπής για το πακέτο φαρμακευτικών προϊόντων. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Α, πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, οι προτάσεις του φαρμακευτικού πακέτου